Jeśli byście Państwo pozwolili, to byśmy rozpoczęli. Μάλιστα, αν επιτρέπετε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη συνεδρίασή μας πολύ καλά. Με ένα τέταρτο καθυστέρηση κιόλα. Περιμένουμε ένα μέρος των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να προσέλθει ακόμα. Δευτέρα είναι, τι να κάνουμε. Και όλοι έχουν φύγει από τις οικογένειές τους για να προσέλθουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου θα είμαστε και στο διαδίκτυο με τη συνεδρίασή μας. Έχουμε διερμηνία σε σχεδόν όλες τις γλώσσες με εξαίρεση τα μαλτέζικα, τα σλοβακικά, τα ε, εστονικά και δεν καταφέραμε να συναντήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα. Αυτό βέβαια συναρτάται και με την κατάσταση της υγείας του Επιτρόπου, αφορά την ίδια την υγεία του. Θα μπορούσε να είχε αντικατασταθεί από τον κύριο Κατάινεν όμως, κατά το πρώτο μέρος της συνάντησης και κατά το δεύτερο από τον Γενικό Διευθυντή Πλέβα, μετά από τη συζήτηση με τους συντονιστές, η πλειοψηφία ε, τοποθετήθηκε υπέρ του να μπορούσαμε ίσως καλύτερα να αναμέναμε να έχουμε μια συζήτηση με τον ίδιο τον Επίτροπο Χόγκαν και όχι με κάποιους αναπληρωτές. Και αυτό τηρήσαμε, αυτό έγινε. Υπήρξαν δύο εναλλακτικές ε, να αναβληθεί για την μηνιολομέλεια, πρώτη εναλλακτική. Δεύτερον, να αναβληθεί για την επόμενη πέμπτη η συνάντηση αυτή. Η γραμματεία ασχολήθηκε με το θέμα και απέρευσε μετά από αυτή την ενασχόληση ότι ήμασταν υπέρ της μηνιολομέλειας ως χρονική στιγμής για αυτή τη συνάντηση. Και ήταν και η βούληση εξάλλου της πλειοψηφίας. Δεν έχουμε ακόμα κάποια συγκεκριμένη, κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά περίπου γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της μήλιολομέλειας θα το έχουμε. Με διορθώνουν, μόλις με διόρθωσαν. Γύρω στις 7 η ώρα το απόγευμα, 19.00 και θα πρέπει ακριβώς να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η μερίσια διάταξη σε σχέση με τις 19.00 ή 20.00. Σημαντικό είναι να γίνει κατά την Ολομέλεια, μην η Ολομέλεια των Βρυξελών. Πρόκειται λοιπόν για την κρίση στον γεωργικό τομέα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σχετικά ότι σήμερα και αύριο το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ε, συναντάτε στο Λουξεμβούργο και γνωρίζετε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με τις ποσοστώσεις και το τι συμβαίνει σχετικά και σε σχέση με τον προϋπολογισμό για την γεωργία και την, ε, τις εξαιρέσεις ή συμπερίληψη ή αν από το αποθεματικό θα καλυφθούν δαπάνες. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα αποτελέσουν θέμα αυτών των διαβουλεύσεων της Συνόδου των Υπουργών Γεωργίας. Και φυσικά θα πρέπει να συζητηθούν και οι αρχές, οι ρήτρες σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη-μέλη μπορούν να δράσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Αυτές είναι λοιπόν γενικές πληροφορίες μετά από την συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας θα γνωρίζουμε φυσικά περισσότερα και τότε θα, μπορούς, μπορέσουμε φυσικά να θέσουμε και ερωτήσεις στον ίδιο τον Επίτροπο την Τετάρτη. Αυτά για αυτό το θέμα. Και <clears throat> γνωρίζοντας τα σχετικά σε σχέση με τις θερινές διακοπές είχαμε επαφές και ανταλλάξαμε απόψεις διότι είναι γνωστό κατά τα άλλα ότι είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. Συναντήσαμε γεωργούς, συναντήσαμε εκπροσώπους του γεωργικού τομέα κατά τις επαφές αυτές και όλοι βρισκόμαστε υπό πίεση, υπό συγκεκριμένη πίεση. Έπρεπε να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις γεωργών για να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα. Και είναι φυσικά σημαντικό να μπορούμε να δίνουμε, να ενημερώνουμε σχετικά. Αυτά σε σχέση με αυτό το θέμα. Περνάμε στο επόμενο, αν δεν υπάρχουν βέβαια κάποιες ερωτήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρεμβάσεις ή ερωτήσεις και περνάμε στο σημείο 3. Τη ημερήσιας διάταξής μας που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 15ης και 16ης Ιουλίου 2015. Θα κάνουμε αυτό το οποίο ήθιστε να γίνεται. Όπως ε, πάντα, αν μέχρι το τέλος δεν υπάρξουν κάποιες ενστάσεις θα θεωρηθεί ότι κυρώνονται. Έχω και μια συγκεκριμένη ξεχωριστή πληροφορία ίσως ε, σε σχέση με αυτό το θέμα θα πρέπει να το εξετάσουμε είναι η συνεδρίαση κατά την οποία η κυρία Πόλσεν που έκανε τόσα πολλά για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και για την ε, Επιτροπή Γεωργίας και για τους γεωργούς που κατέβαλε τόσες προσπάθειες για τα θέματά μας ε, τα οποία ιδιαίτερα αφορούν την υγεία των ζώων και άλλα πολλά σχηδή θέματα είναι ένα άτομο που μπορεί κανείς να βασίζεται πάντα σε αυτό και στις απόψεις και τις δράσεις του. Και τι έγινε ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα είχε εκπονήσει και είχε εργαστεί επ' αυτόν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Και ευχόμαστε όλα τα καλά στην κυρία Όλσεν και λέμε επίσης ότι όλα αυτά τα θέματα που κατά το παρελθόν εκπονήθηκαν, που είχε αναλάβει και εξεπώνησε, ελπίζουμε ότι θα είναι δυνατόν αν υπάρχουν ερωτήσεις να στραφούμε προς απάντηση ερωτήσεων ή παρεμβάσεων για τα συναφή αυτά θέματα και ελπίζουμε ότι θα βασιζόμαστε, θα μπορούμε να βασιστούμε στη δική της, στις γνώσεις της και στην τεχνογνωσία της στο μέλλον. Θα είναι φυσικά πολύ καλό στο μέλλον, πολύ θετικό για μας να μπορούσαμε να την χαιρετήσουμε κατά τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής με ενδεχόμενη συμμετοχή από πλευράς της. Αυτά είχα να σας πω. Θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες και θέλω να σας ευχηθώ όλα τα καλά αγαπητοί για το επόμενο αυτό, την επόμενη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. Και αν θέλετε να πείτε δύο λόγια, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση μπορώ να πω ότι παρακολούθησα και συμμετείχα, με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα και εργαζόμουνα και ήταν η πρώτη θέση την οποία απέκτησα και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου ε, συνέγραψα και βιβλία και μελέτες και γι' αυτό, ήταν για μένα ένα ιδιαίτερα θετικό βίωμα και τώρα μπορώ να πηγαίνω στην Ισπανία, στην Ιταλία και ε, σε σχέση με τον σύζυγό μου και την ε, κοινή μας ζωή νομίζω ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα θετικό. Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να θυμόσαστε ότι αφενός χρειάζονται οι άνθρωποι τρόφιμα για τις επισητιστικές τους ανάγκες. Χρειαζόμαστε τους χώρους της υπαίθρου που πρέπει να, είναι, να μπορούν να λειτουργούν σωστά και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι και η βιολογική οι όροι, προϋποθέσεις και οικονομικοί και όλες οι πτυχές που αφορούν τη γεωργία πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη επαρκώς και να καλύπτονται. Και ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών ζουν πλέον σε αστικά κέντρα, σε πόλεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουν ζωντανά τα χωριά για να είναι ζωντανή η ύπεθρος και να μπορέσει να επιβιώσει και πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων της υγείας των ε, δραστηριοτήτων της γεωργίας καθώς επίσης και των κλιματικών θεμάτων. Όλα αυτά συναρτώνται και συνδέονται πολύ στενά. Παρακαλώ το σύνολο αυτών των θεμάτων να το λαμβάνετε πάντα ολιστικά, σφαιρικά υπόψη και να καταβάλλετε προσπάθειες για το χώρο της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε και πάλι για αυτά τα οποία μας είπατε, για τις συμβουλές που μας δώσατε. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία. Η επισητιστική ασφάλεια, η ασφάλεια τροφίμων. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας εύχομαι κάθε καλό και κάθε επιτυχία. θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην Επιτροπή Γεωργίας ανάμεσά μας και ελπίζω ότι θα είναι δυνατόν σύντομα να ε, ακολουθήσει μία πρόσκληση ώστε πριν από τα Χριστούγεννα να μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε ε, θα ήταν κάτι θετικό αυτό με τις καλύτερες ευχές μας λοιπόν και από πλευράς του συντονιστή που το όνομά του από πλευρά του ΕΛΚ δεν το θυμάμαι. Βοηθήστε με ποιο ήταν το όνομά του. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ και στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Ναι, θα επανέλθει αυτό σε ένα δευτερόλεπτο θα το έχουμε αυτό. Λοιπόν, και παρακαλώ. Ε, ε, ε, αυτό ήταν και σε σχέση με τα θέματα της νοσταλγίας που μας απασχόλησαν περνάμε στο επόμενο σας ευχαριστούμε είναι το 4 η παρουσίαση της έκθεσης της αποστολής αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας Επιτροπής Γεωργίας στις Γαλλικές Άλπεις στην Σαβοία και Άνω Σαβοία αυτές τις περιφέρειες ε, της ε, ε, επαρχίες της Γαλλίας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι φυσικά σε σχέση με τις πληροφορίες έχουμε και το κείμενο στα χέρια μας αλλά δεν είμαι εγώ ο οποίος θα παρουσιάσω το κείμενο της αποστολής αυτής. Είναι ένα, μια εξαιρετική αποστολή, ένα κείμενο που συνοδεύεται από εξαιρετικές φωτογραφίες και ζηλεύει κανείς καμιά φορά βλέποντας ε, αυτά τα τοπία και θα ήθελε κανείς να είχε πάει να πήγαινε ο ίδιος εκεί. Προετοιμάστηκε με εξαιρετικό τρόπο αυτή η αποστολή και στέφτηκε με επιτυχία. Ήταν ιδιαίτερα επιτυχής η αποστολή αυτή. Έχουμε και φωτογραφία των όσων συμμετείχαν. ο κύριος Νταντάν προετοίμασε αυτό το ταξίδι, το διοργάνωσε από υπό κάθε άποψη και σίγουρα κάποιες πληροφορίες θα μπορούσαν να αναφερθούν για αυτή την αποστολή στις Γαλλικές Άλπεις. Διότι επρόκειτο για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες και συναφείς περιφέρειες στην Ευρώπη, ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και πρέπει να αναζητηθούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Κύριε Νταντάν, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ήμουν πολύ ευτυχής που υποδέχτηκα μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην περιοχή μου. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που θέλησα να κάνω είναι να συνδέσω τους αγρότες τους ορεινούς με τα προϊόντα ποιότητας. Δηλαδή, εδώ και ένα μεγάλο διάστημα η Γαλλία έχει προσπαθήσει να υποστηρίξει το εισόδημα αυτών των αγροτών προσπαθώντας να αξιοποιήσει την ποιότητα αυτών των προϊόντων. Είναι pop και τα λοιπά. Έχουμε διαπιστώσει την πρόοδο σε πολλούς τομείς. Το, κράτος, το κρασί, με συγχωρείτε, πρώτα απ' όλα. Ε, και τα πολύ ορεινά τμήματα, φτάσαμε σε πάνω από 2.000 μέτρα υψόμετρο, έχουμε και άλλες παραγωγές. Δυστυχώς ορισμένοι συνάδελφοι νόμιζαν ότι κάναμε ειδικό πρόγραμμα ε, δοκιμασίας τυριών, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι αυτοί που σας υποδέχτηκαν εντυπωσιάστηκαν από τις γνώσεις των μελών της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Ε, δηλαδή γνωρίζουμε πραγματικά τους φακέλους στον τομέα της γεωργίας. Ως προς εσάς κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ να επαναλάβω την επίσκεψη και να σας κάνω ένα θαυμάσιο γύρο του χρόνου στην ίδια περιοχή μου. E, σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω πολύ θερμά να ευχαριστήσω τον Μισελ για την πολύ θετική διοργάνωση αυτής της αποστολής και για τα θέματα για την Επιτροπή Γεωργίας που από πλευρά της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προετοιμάστηκαν πολύ σωστά. Με μεγάλη χαρά γνωρίσαμε αυτές τις περιοχές και διαπιστώσαμε ότι παντού στις Άλπεις τα προβλήματα είναι παρόμοια Ουσιαστικά οι γεωργοί στις ορεινές περιοχές μπορούν να επιβιώσουν μόνο με ποιοτικά προϊόντα, με προστατευόμενη προέλευση και διασφάλιση της προέλευσης αυτής και αυτό εξόφθαλμα καταδείχθηκε. Είδαμε και τις διαφορές που υπάρχουν και τι μπορεί να συμβεί αν δεν διασφαλίζεται η διαδοχή στις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και δεν πιστούν οι νέοι να ασχοληθούν με αυτές τις δραστηριότητες. Τότε παραμένουν χέρσες ακαλλιέργητες ε, και παραμένουν ε, οι ανεκμετάλλευτες, οι περιοχές που είναι τόσο σημαντικές και υπάρχει η δυνατότητα από την άλλη πλευρά παρακολούθησης αθλημάτων χειμερινών όπως σκι ε, όσον αφορά και το κρασί το οποίο μπορέσαμε να δοκιμάσουμε, σε ευχαριστούμε Μισελ Νταντά για τις προσπάθειες που κατέβα. Πρόεδρος, τώρα ζηλεύω ακόμη παραπάνω. Ο κύριος Παζόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πράγματι υπάρχει κίνδυνος ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο του περιφήμου πλαισίου των προελεύσεων διότι τα θέματα δεν είναι σαφή. Όσον αφορά την ανισαβοία το ποσό που πληρω... καταβάλλεται στους αγρότες είναι οπωσδήποτε υψηλότερο αλλά και το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι οι αγρότες της περιοχής πραγματικά ανησυχούν με την εξέλιξη των τιμών. Ευχαριστούμε κυρία Σόντρα. Ε, Μάλιστα και εγώ πήγα σε αυτή την αποστολή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μισελ για την υποδοχή και για την διοργάνωση αυτών των συναντήσεων. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσω να δω και να αξιολογήσω το τι συνεισφέρει που είναι τόσο σημαντικό η δραστηριότητα αυτή, η άμεση πώληση για να μπορούν να διασφαλίζονται τα εισοδήματα των γεωργών. Στην ε, εργασία προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να κάνει πολλά περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαταλείπει στην τύχη τους ε, αυτούς τους παραγωγούς ε, που επιλέγουν την άμεση πώληση γενικά και νομίζω ότι από την Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να κάνουμε σημαντική φανταστικό έργο σε πολλούς τομείς. Ένα, όλες οι όλοι οι τομείς οι φυτοϊγειονομικοί και οι υγειονομικοί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μικρών εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται με τις άμεσες πωλήσει. Δεύτερον, η επίσκεψη ήταν πολύ σημαντική να δούμε το ρόλο των μικρών εκμεταλλεύσεων για τη δραστηριότητα στην παραγωγή στις ορεινές ζώνες και ιδιαίτερα στα ψηλά βουνά, στις υψηλές ορεινές ζώνες. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλές ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να, με αυτή την παρουσία να υποστηρίξουμε τους γεωργούς και κτηνοτρόφους στην παρουσία τους στις ορεινές ζώνες. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η αποστολή, αυτή η επίσκεψη για μένα. Επαναλαμβάνω, έχουμε ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να υποστηρίξουμε και να προαγάγουμε την ορεινή γεωργία και τις άμεσες πωλήσει. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για τη διοργάνωση αυτής της αποστολής, αυτής Πρόεδρο, σα Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συμφωνούμε όλοι να απευθύνουμε ευχαριστίες και θα ήθελα να υπογραμμίσω ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό είναι το θέμα το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε. Είναι πολύ ποικιλόμορφη η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Συνεπώς έχουμε και αυτό είναι θετικό, πολλούς μηχανισμούς μέσα στην κοινή αγροτική πολιτική μας. Έχουμε άμεσες πωλήσει, έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις, αλλά ασχολούμεθα και με τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, με υψηλό κόστος που αντιμετωπίζουν ειδικέ περιστάσεις. Και βεβαίως και τα η προστατευόμενη προέλευση είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευαίσθητα είναι όλα αυτά τα θέματα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που θα ενταχθούν στις όλες τις διεργασίες της Επιτροπής μας και θα μπορέσουμε αυτά τα συμπεράσματα να τα περάσουμε και στην Κομισιόν. Τέτοιες αποστολές είναι πολύ χρήσιμες και θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Πάμε τώρα στο 5 σας παρακαλώ. Παρουσίαση από την εισηγήτρια σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Η εισηγήτριά μας είναι η κυρία Μάκεντάιρ. Θα συζητήσουμε την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς για τα φυτά. Ε, αυτή η πρόταση συζητιέται από το Συμβουλίο εδώ και ένα χρόνο. Τον Απρίλιο του 2014 είχε τοποθετηθεί ήδη το Κοινοβούλιο με την προηγούμενη θητεία του, αλλά το θέμα ήταν αμφισβητούμενο στο Συμβούλιο και το Κορεπέρ υιοθέτησε τέλο πάντων μία θέση 30 Ιουνίου. Στο Σεπτέμβριο του 2014 η Επιτροπή μας είχε ταχθεί με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ μιας, της έναρξης ε, διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Φάιμεν ήταν ε, ο αρχικός εισηγητής, ε, δεν επανεξελέγει και ανέλαβε η κυρία Μάκεντάιρ. Η κυρία Μαρκαντάιρ έχει ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται τις διεργασίες σε σχέση με αυτή την έκθεση και ήδη είχαν μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο σχετικά και είχαμε 136 τροπολογίες στην πρώτη ανάγνωση, αν θυμόσαστε. Τώρα αυτά συζητούνται από το Συμβούλιο των Υπουργών η πρώτη τριμερή συζήτηση θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου. Ε, κυρία Μακεντάιρ, έχετε τώρα το λόγο για να μας ενημερώσετε σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά αυτόν τον πολύ σημαντικό φάκελο. Πώς έχουν τα πράγματα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ σωστή σύνοψη της κατάστασης. Ε, συγγνώμη συνάδελφοι αν θα επαναλάβω κάτι που είπε ήδη ο Πρόεδρος. Όλα αυτά ξεκίνησαν λοιπόν με μία αξιολόγηση των σημερινών κανόνων των ε, φυτο, των για τα φυτά δηλαδή γιατί τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε δει πολλές επιδημίες στα εσπεριδοειδή ε, και σε άλλα δέντρα τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλα κόστη όσον αφορά την ανεπαρκή συνεπώς προστασία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση το 2010 αντιμετωπίσαμε, διαπιστώσαμε μάλλον ότι δεν υπάρχει αρκετή πρόληψη όσον αφορά τις εισαγωγές υψηλού κινδύνου. Επίσης, Υπάρχει, ε, πρέπει να ασχοληθούμε με τη μη εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε δηλαδή πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την, τον έλεγχο της μη εξάπλωσης. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε επίσης τους μηχανισμούς ενδοκινοτικών μεταφορών και προστατευόμενων ζωνών. Η Κομισιόν λοιπόν υπέβαλε ένα νέο σχέδιο κανονισμού τον Μάιο του 2013 για να αντικαταστήσει την υφιστάμενη οδηγία και να επικαιροποιήσει το καθεστώς. Όπως μας είπε ήδη ο Πρόεδρος, η Επιτροπή Γεωργίας υιοθέτησε, ενέκρινε την έκθεση του συναδέλφου Φάινμαν για τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 2014. Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2014 και έτυχε μεγάλης πλειοψηφίας. 476 υπέρ νομίζω ψήφους είχε. Υπογραμμίσαμε λοιπόν τα μέτρα πρόληψης και της πρόορης ανείχνευσης των επιβλαβών οργανισμών. Μετά τις εκλογές εξετάσαμε και πάλι την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή μας λοιπόν ενέκρινε αυτή την εντολή τον Σεπτεμβρίο του 2014. Το Συμβούλιο κατέληξε σε μία θέση τον Ιούλιο του 2015 και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ε, τριμερή διαπραγμάτευση. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου. Θα γίνει μία προπαρασκευαστική συνάντηση βέβαια για να συζητήσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου εν λεπτομερία. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση των ε, σκιωδών εκπροσώπων, διότι ορισμένοι αντιπρόσωποι είναι πολύ καινούργοι αν θέλετε σε σχέση με αυτό το φάκελο. Θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τις απόψεις τους όσον αφορά τις τροπολογίες. Υπάρχουν ε, πολλά θέματα στα οποία το Συμβουλίο, για τα οποία το Συμβουλίο έχει ε, προτείνει μεγάλες αλλαγές. Εν ώψη αυτού ζήτησα λοιπόν από το Συμβούλιο και την Κομισιό να κάνουν μια νική περιουσίαση της θέσης του στην πρώτη παρασκευαστική συνάντηση που θα έχουμε στις 22 Οκτωβρίου. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή των μελών σε ορισμένου τομεί όπου υπάρχει πραγματική διαφορά μεταξύ Συμβουλίου και ε, Κοινοβουλίου. Πρόκειται για τη χρήση της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη θέλουν εφαρμοστικές πράξεις και όχι κατεξουσιοδότηση πράξεις που εμείς προτιμούμε. Επίσης υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το καθεστώς εισαγωγής των φυτών. Η πρόταση του Συμβουλίου δεν είναι σαφής και πιστεύω ότι είναι, αν θέλετε, το πιο δύσκολο θέμα προς διαπραγμάτευση τις επόμενες εβδομάδες. Κατά την άποψή μου, ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει μια ισορροπημένη θέση, να ενισχύσουμε τη σημερινή κατάσταση και να είμαστε ε, σαφείς όσον αφορά ε, τα, τους επιβλαβείς οργανισμούς χωρίς να προσθέτουμε πρόσθετα βάρη στη βιομηχανία ή στις αρμόδιες αρχές. Συνεπώς, θέλω με τους άλλους εκπροσώπους του Σκιώδης να συνεργαστώ πολύ στενά και θα σας αναφέρουμε τα αποτελέσματα στην Επιτροπή μελλοντικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και ζητώ συγγνώμη ε, να σας ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την ενημέρωση και να δώσω το λόγο στον κύριο Χάιταμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους και την κυρία Μάκεντάερ. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχαμε πολύ καλή αρχή, πολλά υποσχόμενη, ε, γιατί το θέμα είναι και καινοτόμο αλλά και πολύ ευρύ, καλύπτει ε, άπτεται πολλών ε, άλλων πτυχών. Είναι σημαντικέ λοιπόν οι αποφάσει που θα πάρουμε εδώ και πρέπει να δούμε ο κλάδο αυτό τι σημασία έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θέλουμε να καλύψουμε υπολογίζουμε σε 30 δις ευρώ ετησίως τον ε, κύκλο εργασιών ε, για τα φυτικά προϊόντα με πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης. Οπότε οι αποφάσεις που θα βάλουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να φροντίσουμε να διαφυλάξουμε ότι υπάρχει, διότι το σύστημα αυτό υπάρχει από το 1977 κοινό κρεβονίο λίθος για την προστασία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, χωρίς όμως να εμποδίζουμε τις εμπορικές ροές και την οικονομική ανάπτυξη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το σύστημα αυτό. Γι' αυτό και το Ευρωκοινοβούλιο ήδη σε δύο διαφορετικέ περιστάσει έχει αποφασίσει ότι το σύστημα αυτό είναι καθοριστική σημασία για όλε τι εμπορικέ μα συναλλαγέ. Κατά πρώτον, λοιπόν, όπω ανέφερε και η κυρία Μάκινταερ και στην ε, Σύνοδο τη Ολομέλεια τον Απρίλιο του 2014, με τι τροπολογίε για το άρθρο 40 που πρότειναν ένα κλειστό σύστημα, είχαμε την ε, απόρρεψή τους κατά συντριπτική πλειοψηφία. Και ε, στην, ε, στο ψήφισμα για την Ψιλέλα στην Νοτοιταλία και εκεί οι σχετικές τροπολογίες απορρίφθηκαν. το κλειστό σύστημα θα εμπόδιζε το ελεύθερο εμπόριο και θα χάναμε θέσεις εργασίας και καινοτομία με τη δημιουργία συγκεκριμένων θυλάκων εμπορικών ε, θα χάναν 4 δις ευρώ οι Ευρωπαίοι Γεωργοί. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η αντίδραση ε, είναι ε, σημαντική. Εδώ εάν εφαρμόζαμε ένα κλειστό σύστημα και οι τρίτες χώρες γύρω μας θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και να βλάψουν το εμπόριο ακόμη περισσότερο. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε, να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο κλειστό σύστημα θα πρέπει να έχουμε μια μελέτη αντικτύπου για να το πράξουμε. Διότι οι οικονομικές συνέπειες δεν μπορούν να παραπλευτούν. Εάν θέλουμε τέτοια μελέτη αντικτή που μπορεί να εκπονηθεί, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον μια διετία και αυτό θα καθυστερήσει πολύ την περαιτέρω επεξεργασία τη πρόταση. Για να ολοκληρώσω, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό το σύστημα, το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φυτικά προϊόντα και δεν θέλουμε ένα κλειστό σύστημα που θα το εμπόδισε. Ε, πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο με την Επιτροπή Γεωργία να δώσει μια ισχυρή εντολή στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο για να διαφυλάξουμε το ανοιχτό σύστημα και να είμαστε σταθεροί στι απόψει μα. Να μην δεχτούμε το άρθρο 41α τη τωρινή πρόταση που ε, εισάγει ένα νέο σύστημα το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με ένα σύστημα που θα ήταν κλειστό. Ευχαριστώ κυρία Σνάγερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το είδαμε αυτό σε σχέση με την τήρηση των φυτογειονομικών διατάξεων. Εδώ σε σχέση με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για ειδική προστασία που την χάνει η συζήτηση στην Ολλανδία πρέπει οι ζώνες αυτές να καθοριστούν και να ε, χρησιμοποιούμε καλύτερα τους ε, κανόνες αυτούς. Αυτό ισχύει για αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει και οι επιχειρηματίες να εμπλέκονται ώστε στο σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σημερινό σύστημα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανατραπεί. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν προβλήματα στην αγορά επιβάλλοντας κάποιες διατάξεις ή τροχοπεδώντας κάποιες άλλες. Πέρυσι είδαμε τη δυνατότητα θετικών συνδυασμών της ελευθερίας, της ελεύθερης αγοράς με τις ενδεδειγμένες αυτές δράσεις της το υγειονομικές, ώστε να υπάρξει ένα παγιωμένο σύστημα. Όμως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει για να το πετύχει. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και τώρα η κυρία Αγγιλάρ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ από πλευράς μου παρότι δεν ε, παρακολούθησα και δεν βίωσα την έγκριση αυτής της εντολής, θα ήθελα να δραχθώ της ευκαιρίας να τονίσω κάτι, να τονίσω την εντύπωση που έχω αποκομίσει για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό και κατανοώ βέβαια το θέμα, την θέση των φιλελεύθερων. Όμως το σύστημα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Οι έλεγχοι στα σύνορα δεν λειτουργούν έχουμε μια εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια συγκεκριμένη πανόλης ε, παρασίτων που πλήττουν ιδιαίτερα τις χώρες της Μεσογείου επειδή δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος των συνόρων της Ευρώπης και είναι μια πραγματική κατάσταση αυτή, ένα δεδομένο και πιστεύω ότι αναφερόμενοι σε σχέση με αυτό, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό βέβαια το ελεύθερο εμπόριο. Είναι πολύ σημαντικό. Όμως και η έλεγχη στα σύνορα είναι πολύ σημαντική να πρέπει να πληρώνουν οι παραγωγοί ή να πληρώνουν οι καταναλωτές για τέτοιου είδους ε, όπως για παράδειγμα την, ε, ε, τις μελανές κοιλίδες ή την, τα παράσιτα αυτά της πανόλης αυτής δεν είναι λογικό. Κάτι πρέπει να γίνει και το θέμα πρέπει να διευθετηθεί και πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να μείνουμε ε, τροχοπεδημένοι και ακίνητοι λόγω του Συμβουλίου. Είναι αναγκαίο να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν λειτουργούν καλά αυτή τη στιγμή. Και οι κυριότεροι οι οποίοι επιζημιώνονται ε, σήμερα είναι οι Ευρωπαίοι παραγωγή. η ευρωπαϊκή παραγωγή. Και σε σχέση με το σημερινό σύστημα πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει, να τροποποιηθεί. Πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις και φυσικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγμα που είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δράσουμε για να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ντομάτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να συνεισφέρω στην συζήτηση. Έστω και τώρα, γιατί δεν είχα διαβάσει το σχέδιο κανονισμού για τα φυγειονομικά μέτρα για τους επικλαβούς οργανισμούς στα φυτά. Είναι σημαντικό επειδή θα είμαι και όντως εισηγήτρια στους επόμενους τρομερεί διαλόγους. Ασχολούμαι εδώ και μήνε με το πρόβλημα της ξηρέλαφας στην Διόζα που όλοι γνωρίζετε πολύ καλά και είδα από κοντά τις σοβαράτατες συνέπειες από λανθασμένες ε, λύσεις που βρέθηκαν ως τώρα για το πρόβλημα αυτό και ότι ζημιά μπορεί να προκαλέσουν στη γεωργία μας και την οικονομία μας. Γι' αυτό έχω την πρόθεση στους τριμερείς διαλόγους να στηρίξω όλα τα μέτρα που αφορούν την πρόληψη και την πρόορη διάγνωση των παθογόνων οργανισμών όλοι οι οργανισμοί που θα έπρεπε να βρίσκονται σε καραντίνα και που επιτίθενται στα, είναι επιβλαβείς για τα φυτά θα πρέπει να προστατεύονται με κάθε τρόπο, ε, από κάθε, με κάθε γνώση της βιοπονικής που διαθέτουμε και στην πράξη. Θα πρέπει τα φυγειονομικά μέτρα να είναι η τελευταία μας λύση και να δίδεται ε, προτεραιότητα στις ουσίες που επιτρέπονται στην βιολογική γεωργία ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη βιολογική ασφάλεια με τις απαραίτητες οικονομικές ε, εξισορροπήσεις για τους γεωργούς. Επίσης, ο κατάλογος για τους επιπλαβείς οργανισμούς ε, κατά των φυτών κατάλογος που ως τώρα έχει εκπονηθεί θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να συμπεριλάβει και άλλους οργανισμούς. Για την ε, εκρίζωση του βακτηριδίου της κλειολαφαστιδιόζα λόγου χάρη στην Απουλία δεν είναι το ίδιο που θα χρειαζόταν να κάνουμε και με τα ίδια μέτρα στην Κορσική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις των βακτηριδίων ε, σε κάθε περίπτωση και το πώς οι επιβλαβείς οργανισμού μπορούν να μεταλλαχθούν. Θα πρέπει αυτούς τους παθογόνους οργανισμούς να το δούμε σε, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τώρα η προσέγγιση μα είναι σαφώ λανθασμένη και καταστρέφουμε τη γεωργία και την οικονομία σε ένα μεγάλο μέρο τη Ένωση. Μέσω τη τελευταία πρόταση τη ε, συναδέλφου Μάκεντάιρ θα πρέπει να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ο κύριος Σεμπάστιαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμμετέχοντας σε αυτό το θέμα δεν ήμουν προηγούμενα Ευρωβουλευτής και έτσι ασχολούμαι τώρα με αυτό. Έχει τεράστια σπουδαιότητα αυτό το οποίο εξετάζουμε, διότι το θέμα των ασθενειών αυτών και των παρασίτων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττει ιδιαίτερα ως μάστιγα τις χώρες του Νότου. Και στη δική μας περιοχή κάθε χρόνο έχουν οι όλο και περισσότερο φόβο ότι οι μαύρες, οι μελανές αυτές κοιλίδες θα πλήξουν τις καλλιέργειες και αυτό το βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, για παράδειγμα για διάφορα πλοία τα οποία έχουν ε, ελεγχθεί στην ε, Βαλένθια και που έχουν υποστεί εμπάργο των φορτίων τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν λειτουργεί το συνολικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Είναι ένα δόγμα το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η κατάσταση. Πρέπει να θυμηθούμε ότι υφιστάμεθα τώρα τώρα τις ε, κλιματικές αλλαγές ήδη σήμερα. Έτσι λοιπόν προσαρμόζονται αυτές ε, οι παρασιτικές ε, καλλιέργειες και έτσι πλήττουν τον νότο της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα κλειστό σύστημα. Παρακολύεται η ελεύθερη κυκλοφορία και μπορεί να έχει πολύ αρνητικέ επιπτώσεις. Αληθεύει ότι ένα αληθινό αληθές ανοιχτό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα με πολύ προβληματικές καταστάσεις. Εμείς είμαστε υπέρ του να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να γίνει για την πρόληψη και να μπορέσουμε με την θέσπιση ενός σαφούς καταλόγου εκείνων των χωρών που είναι ασφαλείς και των άλλων που δεν θα θεωρούνται ασφαλείς ώστε να είναι σαφής η κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεισφέρουμε λοιπόν ώστε αυτός ο κανονισμός να είναι το δυνατόν ο καλύτερος. Και ευχαριστούμε φυσικά για το έργο της εισηγήτριας κυρίας Μακιντάιρ που πολύ καλά έχει διοργανώσει το θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Λοιπόν εγώ δεν θα επαναλάβω τις παρεμβάσεις που έγιναν, την παρέμβαση της κυρίας Αγιούσο που για λόγους ε, που δεν μπορούσε να, μπορούσε να αναβάλει δεν μπορεί να παραστεί και μου ζήτησε να παρέμβω εξ ονόματός της. Ε, και θα ήθελα γι' αυτό πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Μάκιντάε Πρόεδρε για την συνάντηση των σκιωδών ε, εισηγητών που διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα και όπου υπήρχε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις απόψεις που είχαν οι συντονιστές, οι σκιώδεις εισηγητές για αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη εκτίθεται, λέει η κυρία Γιούσο, σε μεγάλους κινδύνους φυτοϊγειονομικούς και όταν έχουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα πρέπει να αποφύγουμε νέα προβλήματα να εισέρχονται, να διεισδύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να προστατέψουμε τους παραγωγούς και τον τομέα τους και την παραγωγή τους. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική ελέγχων εισαγωγών που θα είναι αποτελεσματική και θα δώσει τη δυνατότητα αναβάθμισης φυτογειονομικά των διαδικασιών και θα δώσει τη δυνατότητα δυνατότητα να γνωρίζουμε καλύτερα τι γίνεται με τα φυτογενομικά θέματα και τα φυτά που ε, εισέρχονται και εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως αναφέρθηκε εδώ το θέμα της συλλέγια και, ε, που είναι ένα πολύ σημαντικό βακτηρίδιο και που έχει πλήξει ένα σημαντικό, ε, σημαντικότατες καλλιέργειες και στο νότο της Ιταλίας και έχουν οδηγήσει, έχει οδηγήσει η ξυλέλα φαστιδιώσα σε μεγάλες απώλειες στους ελαιώνες της Απουλίας την περασμένη άνοιξη. Και θέλω λοιπόν να το τονίσω αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στην ενισχύη νομοθεσία ώστε να είμαστε πολύ πιο καλά επικεντρωμένοι και εστιασμένοι στην πρόληψη. Πρέπει σε σχέση με τα φυτοκτόνα να, είναι, να δούμε ότι είναι πολύ περιορισμένη η χρήση τους λόγω της αυστηρής νομοθεσίας που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε την ε, ε, ε, ε για τα φυτογενομικά, ιδιαίτερα για τις νέες ασθένειες που αφορούν τρίτες χώρες και που δεν υπάρχουν για αυτές θεραπείες επαρκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άποψή μου είναι, λέει η κυρία Αγιούσο, ότι η θέση του Συμβουλίου παρουσιάζει κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι μια συμβιβαστική λύση μεταξύ ακραίων θέσεων και τοποθετήσεων. Όμως, σε σχέση με διαφορετικά κεφάλαια του κανονισμού δεν ελήφθησαν υπόψη κάποιε πολύ λογικές στρατηγικές προτάσεις που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως είναι οι διαδικασίες που επιβάλλονται σε σχέση με το διαμετακομιστικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε τη διάδοση, τη διάχυση αυτών των ασθενειών. Επιμένει και μένει η κυρία Αγιούσο ότι πρέπει σε αυτή την επικέντρωση να παραμείνουμε σωστοί σε σχέση με καταλόγους ασθενειών ώστε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε καλύτερη νομική, βελτιωμένη νομική ασφάλεια, καλύτερη νομική βεβαιότητα είναι πεισμένη ότι η κυρία Γιούσο ότι με τη συνεργασία όλων μπορούμε πολύ γοργά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία πολύ σύντομα που είναι για ένα θέμα που είναι τόσο σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Αυτά είχα να πω. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεκάστρο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα μόνο δευτερόλεπτα για να συγχαρώ τη συνάδελφο Μάκινταρ για την εξαιρετική της δουλειά. Αναμφίβολα. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. Με την ανησυχία τους για τα φυτογενομικά μέτρα, για τα φυτά που έχουν πληγεί και γιατί είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια προέκυψαν προβλήματα, όπως με την ξυλέλαφα στην στην περίπτωση αυτή είδαμε ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα. Έχουμε πλέον τη βεβαιότητα ότι τα καλοπιστικά φύτα από την Κωνσταντίνα δημιούργησαν αυτήν την, προκάλεσαν αυτή την επιδημία με όλες τις συνέπειες που ε, όλοι οι συνάδελφοι εντόπισαν. Ε, με όσα λοιπόν ψηφίσαμε, βλέπουμε ότι πρέπει να προβλέψουμε ε, όρια και έλεγχο στις εισαγωγές, γιατί όσα ως τώρα ισχύουν βλέπουμε ότι δεν αρκούν. Δεν θέλουμε να παγκοσμιοποιηθούν και οι επιδημίες ε, στο μέλλον, δημιουργώντας ακόμη σοβαρότερα προβλήματα για τους γεωργούς μας. Έχουμε εξαντλήσει το κατάλογο των ομιλητών, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συγκήτριά μας για να σχολιάσει όσα ελέγχθησαν. Η κυρία Μακεντάιρα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες επειδή δια αν τις απόψεις του σήμερα. Δεν θα ήθελα να απαντήσω ή να σχολιάσω όσα ελέγχθησαν. Τα έχω όλα σημειώσει λεπτομερώς και πιστεύω <clears throat> ότι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια ισορροπημένη θέση και τοποθέτηση και αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εξή ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού σχετικά με τη σφαγή ζώων. Στην συνάντηση των συντονιστών 5 Μαΐου και μετά από πρόταση που έγινε, οι συντονιστές αποφάσισαν να θέσουν το θέμα της τελετουργικής φαγής και να το συμπεριλάβουν στην ημερήσια διάταξη μια συνάντηση της Επιτροπής μας. Τον Ιούλιο λοιπόν συζητήθηκε η πρόταση αυτή με τους συντονιστές, η γραμματεία αποφάσισε να οργανώσει επαφές με πολιτικές ομάδες ώστε να αποφασιστεί το σχήμα της συζήτησης. Η απόφαση των πολιτικών ομάδων ήταν να καλέσουμε έναν ειδικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι σε θέση να αποσαφηνίσει και να μας εξηγήσει τον κανονισμό αυτό τα μέλη της Επιτροπής μας έχουν μεγάλες προσδοκίες για τη σημερινή συζήτηση. Το περιεχόμενο θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα τα οποία θα πραγματοποιήσουμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν αμέσως να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, στον κύριο Ανδρέα Γκαμπινέλη από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Είμαι υπεύθυνο ο Διευθυντής της Υπηρεσίας για, την ε, ζωική, για τα ζωικά προϊόντα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση για την Επιστηστική Ασφάλεια και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Έχουμε μια σύντομη παρουσίαση με κάποια στοιχεία που ελπίζουμε να λειτουργήσει το σύστημα για να τη δούμε. Η παρουσίασή μου σε λίγα λεπτά θέλει να σας παρουσιάσει το πλαίσιο των όσων ισχύουν για τις δραστηριότητες των 100 μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να ελοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένας κανονισμός που επέτρεψε να εξυγχρονιστεί το σύστημα της φαγής των ζώων και να προβλεφθούν προϋποθέσεις για τη ζωική προστασία που βελτιώνουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται και μειώνουν τον πόνο των ζώων. Όσο, από όσα γνωρίζετε, μιλάμε για μια 25.000 βοηθοί που σφαγιάζονται θυσίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, εκατοντάδες χιλιάδες χείρους και ε, πουλερικών είναι ένας κλάδος λοιπόν της οικονομίας με πάρα πολύ σοβαρό ειδικό βάρος. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αλλάξω τη διαφάνεια, ε, προβλέφθηκε και χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με νέα στοιχεία ως προς την ε, παρακολούθηση των διαδικασιών για την αναισθησία με έναν υπάλληλο υπεύθυνο για όλη τη διαδικασία της ζωικής ευζοίας ε, εγκατάσταση και με προϋποθέσεις για τις αρμοδιότητες όλων όλου του προσωπικού που ασχολείται με τα ζώα και έρχεται σε επαφή με αυτά. Ως σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το πλαίσιο για τους ε, ελέγχους και την παρακολούθηση που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλύψει περίπου το 70% των δραστηριοτήτων της Ευρώπης. Χάρη στον κτηνιατρικό οργανισμό έχουμε επισκεφτεί 13 κρατημέλη με πλήρη συνολικό έλεγχο και επειδή οι έλεγχοι εκπονήθηκαν από τους ίδιους υπαλλήλους που ασχολούνται και με τα στοιχεία ασφάλειας των τροφίμων είναι κάτι που μας επιτρέψε να εξοικονομήσουμε πόρους. Και μπορέσαμε και να εκπονήσουμε κάποιες μελέτες ε, μελέτες με στοιχεία οι οποίες μπόρεσαν να αποσταλούν στους αρμόδιους υπαλλήλους. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ έχουμε ένα σύντομο κατάλογο των κρατών που επισκεφθήκαμε για να ενημερωθείτε. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν και κράτη με παραγωγή ιδιαίτερα σοβαρή όπως οι κατοχώρες, η Γερμανία, η Γερμανία και η Γαλλία αλλά και μικρότερες χώρες. Έτσι θελήσαμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος της φαγή ζώων στην Ευρώπη. Μπορούμε να προχωρήσουμε ε, στην καινούργια διαφάνεια. Τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν. Καταρχάς, ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι χάρη στην καλή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, δηλαδή των εκπροσώπων του κλάδου, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, και σε ό,τι αφορά το τεχνικό τμήμα των εμπειρογνωμόνων για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην σφαγή ο κανονισμός έφτασε ένα επίπεδο υλοποίησης πολύ ικανοποιητικό σχεδόν σε όλους τους τομείς. Όλος ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά το κόκκινο κρέας. Απομένει η δυνατότητα να υπάρξουν τεχνικές βελτιώσεις βεβαίως, ιδίως ό,τι αφορά την αναισθησία, την αναισθητοποίηση Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε πώς χρειαστούν και περισσότεροι πόροι. Ο υπεύθυνο ζωικής ευζωίας έχει γίνει πλέον ένα πρόσωπο που είναι αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας ε, ενός φαγείου και επιτρέπει τη βελτίωση των δραστηριοτήτων όλου του κλάδου δίνοντας και τις απαραίτητες εγγύσεις. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε εργαστεί και σε διεθνές επίπεδο για τα θέματα αυτά, όχι μόνο με αυτές με τις διάφορες δημοσίευσεις μας, αλλά και με μια διεθνή διάσκεψη που επέτρεψε να ε, συμμετάσχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και άλλοι ενδιαφερόμενοι και συμμετέχοντες στον κλάδο, ενώ ταυτόχρονα χάρη και στη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το λεγόμενο EU WellNet, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2013 και έδωσε ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την δυνατότητα διάδοσης των καλών πρακτικών πολύ γρήγορα στους αρμόδιους ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με νέες τεχνολογίες που θα επιτρέψουν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι τεχνικές σφαγής. Επόμενη διαφάνεια το εξώφυλλο του φυλαδίου μας, της μπροσούρας μας που έχουμε διαθέσιμη στον ιστότοπο σε διάφορες γλώσσες και σε αντίτυπα που μπορούν να διατεθούν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συνεχίζουμε. Η εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας των ζώων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και το έχουμε ακούσει επανειλημμένος αυτό. Έτσι θα ε, βελτιωθούν οι τεχνικές σφαγής και θα μειωθεί ο πόνος των ζωών. Πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται χωρίς ε, παρέμβαση τρίτων. Γι' αυτό χρειάζεται να δοθεί ε, έμφαση και στο πρόγραμμα καλύτερη εκπαίδευση για ασφαλέστερα τρόφιμα. Με την απαραίτητη εκπαίδευση των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους. Μπορέσαμε να καλύψουμε περίπου 300 άτομα που ασχολούνται με τους ελέγχους στα σφαγεία αυτή τη στιγμή, με τις διαδικασίες αυτής εκπαίδευσης και όχι μόνον, διότι όπως τα γνωρίζετε, ο κανονισμός αυτός ισχύει και για τις περιπτώσεις εξαγωγών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το κρέας, όπου χρειάζεται ειδική ε, προετοιμασία και για τους ταινιάτρους που ασχολούνται με το σκέλος των εξαγωγών να προχωρήσουμε, πηγαίνουμε προς το τέλος. Σίγουρα οι επιστημονικές γνώσεις και οι τεχνολογικές είναι δύο σημαντικά στοιχεία που και η αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων φροντίζει με την συνεισφορά της να μας παράσχει. Σε ό,τι αφορά τον, ε, την αναισθητοποίηση, αλλά και σε σημαντικές τομείς πιο δύσκολους όπως η αναστοποίηση των πολιτικών, εδώ κοιτάζουμε το συσχετισμό μεταξύ της αναστοποίηση με ηλεκτρικά μέσα και την ποιότητα του κρέατος που προκύπτει ανάλογα με τη χρήση ή όχι διαφορετικών μέσων. Δηλαδή μας απασχολούν και οικονομικές συνέπειες σε σχέση με το τι γίνεται στην πράξη. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ κάποια κουπιά εργαλείων, όπως λέγεται τα toolbox με χρήσιμες πληροφορίες. Τα ετοίμασε η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Έρχη για την Ασφάλεια των Τροφίμων, διατίθενται στο διαδίκτυο και παρουσιάζουν τεχνικές πρακτικές πληροφορίες για όσους εργάζονται σε σφαγεία στην Ευρώπη και όχι μόνον. Να μπορέσουν δηλαδή να αξιολογήσουν ίδιο το πώς λειτουργεί το σφαγείο τους και το κατά πόσο υλοποιούν σωστά τον κανονισμό. Είναι ένα <clears throat> σύνολο μέσων πρακτικών για τις καλές πρακτικές, για την παρακολούθηση υλοποίηση της νομοθεσίας και για να δούμε πώς λειτουργεί συνολικά το σύστημα. Νομίζω μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια άλλα στοιχεία. Όπως έλεγα το ευρωπαϊκό σύστημα έχει προβληθεί σε διεθνές επίπεδο ώστε ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων ο ΙΕ όπως ε, είναι τα αρχικά του στις ξένες γλώσσες έχει ουσιαστικά υιοθετήσει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων στα σφαγεία με κατευθυντήριες γραμμές. Κατά τον ίδιο τρόπο εκπονήσαμε ελέγχους σε τρίτες χώρες που είναι η βασική εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βεβαιωθούμε ότι προστατεύονται και οι καταναλωτές ε, ως προς την ποιότητα του εισαγόμενου κρέατος. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για πολλές χώρες, όπως λέτε, η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία είναι χώρες σημαντικές για, το, για την ευρωπαϊκή αγορά. από τις χώρες αυτές έρχεται μια σειρά από διαφορετικά προϊόντα και μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τις χώρες αυτές και με συμφωνίες σύνεργασίες για τον τομέα αυτό. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η Επιτροπή εξέδωσε, όπως έλεγε προηγουμένως, μία έκθεση για την αστυνοποίηση των πολιτικών από το Δεκέμβριο του 2013 με τα πιο πρόσφατα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία για να κατευθύνει τις επενδύσεις στα μέτρα βελτίωσης της ανασυντοποίησης των πουλερικών. Όπως είπα, είναι ο τομέας με τα περισσότερα σφάγια ετησίως. Δισεκατομμύρια πολλές φορές. Τον Μάιο του 2015 υπήρξε και μια μελέτη για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την ανασυντοποίηση. Ε, εδώ συμπεριελήφθη η ανεστοποίηση ή μη σε περιπτώσεις σφαγής ε, για θρησκευτικούς λόγους και μετά ε, έγινε και μια μελέτη ε, για μια έκθεση μάλλον για την σφαγή των βοηδών διαντιστροφής δηλαδή την σφαγή τους για θρησκευτικούς σκοπούς η οποία και αυτή δημοσιεύθηκε αναλόγως. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε την πιο πρόσφατη μελέτη του Μαΐου 2015 που καταλήγει ότι για το θέμα αυτό οι περισσότεροι καταναλωτές δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται πάρα πολύ και είχαμε μάλιστα ένα ευρύτατο δείγμα. Δεν είναι πληροφορίες που τους καίνε τους καταναλωτές. Ε, μεταξύ άλλων, δεν δόθηκε καν η εντύπωση σε όσους πήραν μέρος στις συνεντεύξεις αυτές με τους Ευρωπαίου καταναλωτές ότι είναι απαραίτητες αυτές οι πληροφορίες. Αντιθέτως, η μελέτη υπογραμμίζει ότι η σωστή επισήμανση των προϊόντων ε, μια ετικέτα δηλαδή που θα εξηγεί αν υπήρξε ανιστοποίηση ή όχι, αυτό θα μπορούσε μάλιστα να στιγματίσει τα προϊόντα ή να κάνει διακρίσεις ως προς συγκεκριμένα διαιτολόγια που ακολουθούνται ή την ε, συμμετοχή στις θρησκευτικέ ομάδες στον ευρύτερο πληθυσμό. Τελευταία διαφάνεια, τα συμπεράσματα από τα τελευταία χρόνια δράσης μας. Να θυμίσω ότι τέθηκε σε ισχύ το 2013 ο κανονισμός, δηλαδή δύο χρόνια πραγματικής ε, ισχύω. Μεγάλες καινοτομίε σε σχέση με την οδηγία του 1993 ήταν ότι πραγματικά είχαμε μια επανάσταση σαν αυτή του Κοπέρνικου από πολλέ απόψεις, με φοβερέ τεχνικές ε, αλλαγές τεχνολογικές προσαρμογές σε σχέση με την ε, υγεία των ζώων που απαιτήθηκαν ουσιαστικά από τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Από την άλλη δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα ως προς την υλοποίηση του κανονισμού, μόνο κάποιες δυσκολίες όπου μπορούμε με διευθυντικά μέτρα να παρέμβουμε ή με τεχνικές ε, παρεμβάσεις. Και τελευταίο ε, στοιχείο, η συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη ήταν μια συνεργασία που συνεχίζεται αμύωτη και πολλέ φορέ συμπεριλαμβάνει και τρίτε χώρε. Αυτά ήταν τα ε, σύντομα αποτελέσματα τη έκθεση αυτή για την τελευταία διετία υλοποίηση του κανονισμού. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας. Ο κύριος Βοτσιχόσκι έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης που έγινε αυτή η εισαγωγή για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα πρέπει να πω. Που... Ευχαριστώ τον κύριο Γαβινέλη λοιπόν για την παρουσίαση που μας έκανε. Ήμουν εισηγητής για αυτό το κανονισμό το 2009 όταν ε, η πιο ανθρώπινη σφαγή εισήχθη σαν κανόνας ή με την αναισθητοποίηση και όχι μόνο και μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιστάσεις για θρησκευτικούς λόγους ε, επιτρέπεται την εποχή εκείνη η θανάτωση ενός ζώου, η σφαγή ενός ζώου χωρίς αναισθητοποίηση. Αλλά μόνο για θρησκευτικούς λόγους είχε υπάρξει αυτή η εξαίρεση. Η πρακτική όμως, όπως έχουμε δει και όπως παρατηρούμε, είναι διαφορετική. Ιδιαίτερα στις σφαγές για εξαγωγές. Η ανισθητοποίηση δεν χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτή είναι η πιο πρώτη μου αντίρρηση. Γιατί να έχουμε δηλαδή έναν κανόνα ο οποίος να λέει ότι η ανισθητοποίηση απαιτείται εάν είναι ανεκτή ή αν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μία μέθοδος παραγωγής κρέατος χωρίς αναισθητοποίηση για εξαγωγή. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτού του τύπου οι ερμηνείες καθιστούν τον κανόνα της αναισθητοποίησης τελικά χωρίς περιεχόμενο για τα ζώα. Αν αυτό η εξαίρεση αφορούσε μόνο την θρησκευτική εφαρμογή, θα το καταλάβαινα. Προσωπικά βέβαια δεν πιστεύω ότι αυτή η εξαίρεση για, για θρησκευτικούς λόγους πρέπει να ισχύει. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ελευθερίας του θρησκεύματος, του δόγματος. Νομίζω ότι έχουμε ευρωπαϊκές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές μας μας λένε ότι πρέπει να έχουμε μια ανθρώπινη προσέγγιση προς τα ζώα και να τα ταλαιπωρούμε όσο είναι αυτό δυνατόν. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή έπρεπε να υπάρχει εξαίρεση για θρησκευτικούς λόγους ε, πιστεύουμε στην ανθρώπινη προσέγγιση, όχι στην θρησκευτική προσέγγιση. Η θρησκευτική προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τη σφαγή, δεν έχει κανένα χώρο η θρησκεία εκεί μέσα, δεν μιλάμε για α, ναούς, μιλάμε για σφαγεία. Λοιπόν, για μένα αυτή η εξαίρεση είναι πολύ αμφισβητήσιμη. Εν πάση περιπτώσει, έχει εισαχθεί και θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να την εφαρμόζουμε μόνο στις θρησκευτικέ κοινότητες. Δεν βλέπω κανέναν απολύτως λόγο ε, νομικού, ηθικού ε, περιεχομένου να επιτρέπεται αυτή η μέθοδος φαγής στην παραγωγή κρέατος προς εξαγωγή. Διότι αν το επιτρέψουμε αυτό, πιστεύω ειλικρινά ότι οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση χρήσης της, της αναισθητοποίησης ε, δεν θα έχει κανένα νόημα, θα είναι κοινό θέμα. Ε, κύριε Γκαβινέλη, ε, ποια, είναι η κλίμακα σφαγής παραδείγματος χάρη αγελάδων με αναισθητοποίηση και χωρίς αναισθητοποίηση. Πόσες σφάζονται αγελάδες στην Ευρώπη το χρόνο πόσες με αναισθητοποίηση και πόσες χωρίς. Θα ήθελα τα στοιχεία και για τα πουλερικά σας παρακαλώ ώστε να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτών των αριθμών και των θρησκευτικών κοινοτήτων που επικαλούνται αυτή την εξαίρεση. Συνοψίζω για να καταλήξω. Πιστεύω ότι εξετάζοντας τη σημερινή κατάσταση με τους μετανάστες και με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις αρχές μας, το σύστημα των αρχών μας που περιλαμβάνει και το υπογραμμίζω μία ανθρώπινη προσέγγιση και συμπεριφορά προς τα ζώα. Είναι μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς μας αυτό η συμπεριφορά προς τα ζώα. Προσπαθούμε να μην ταλαιπωρήσουμε τα ζώα πέραν ενός σημείου. Χρησιμοποιούμε βεβαίως τα ζώα αλλά με τρόπο που να συνεπάγεται το μικρότερο πόνο ε, εφικτό. Στην ομάδα ευζοίας έχουμε δει πραγματικά μακάβριες ταινίε όσον αφορά τις μεθόδους φαγής. Έχουμε δει πόσο άσχημα υποφέρουν, πόσο πολύ υποφέρουν αυτά τα ζώα και πρέπει πραγματικά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην συμβαίνει αυτό επωνόματι των ευρωπαϊκών μας αρχών. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ μετά από όσα ελέγχθησαν. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Ε, σφαγή χωρίς ε, ανισθητοποίηση για εξαγωγή. Αναφέρεται αυτό στις παραγγελίες για θρησκευτικέ κοινότητες ή να ρωτήσω διαφορετικά, χωρίς αναισθητοποίηση, εξαγωγές, πρόκειται για παραγγελίες από θρησκευτικέ κοινότητες ή γενική πρακτική για τις εξαγωγές. Η κυρία Πόλσεν έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που γίνεται αυτή η συζήτηση Χαίρομαι που υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που εφαρμόζεται από τα σφαγεία, που εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά μας πρότυπα και συμφωνώ με τον κύριο Καλκόψη ότι και εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ τις σφαγές χαλάλ και κόσερ για θρησκευτικούς λόγους. Δεν μπορώ να προσπίσω αυτή την προσέγγιση. Η Ευρώπη είναι χριστιανική περιοχή βασικά. Και αν πάμε τώρα στα αρχικά κείμενα της χριστιανικής μας βίβλου, θα δούμε, και το λέμε αυτό συχνά, ότι παραδείγματο χάρη η ομοφιλοφιλία είναι λάθος, είναι φοβερή, είναι αμαρτία. Λοιπόν, εμείς βέβαια δεν το πιστεύουμε πια αυτό στην Ευρώπη. Δεν το δεχόμαστε αυτό σαν αρχή. Θεωρούμε ότι αποτελεί αντικείμενο της ατομικής ελευθερίας και έχουμε εξίσου καλούς λόγους για να εξετάσουμε και να σκεφτούμε ε, αν πρέπει να μην αναισθητοποιούμε ορισμένα ζώα ή όχι. Κύριε Γκαβινέλη, σας παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε τι ποσοστό των ζώων της Ευρώπης, από όλα τα εκατομμύρια ζώα που σφάζονται, τι ποσοστό σφάζονται χωρίς ανισθητοποίηση. σας παρακαλώ. Πρόεδρος. Πολύ σας ευχαριστούμε. Γνωρίζουμε ότι σε λίγο θα αποχωρήσετε και θα θέλαμε λοιπόν να σας συγχαρούμε με αυτή την ανθοδέσμη. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Πάντα είσαστε ε, και πάντα με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα σας έχουμε ανάμεσά μας. Τώρα έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι απολύτως αναγκαίο και απαραίτητο η χνηλασιμότητα να καθοριστεί με την ε, όσο πιο γίνεται διεξοδική επισήμανση, όχι μόνο για την προέλευση του κρέατο, αλλά και για τον τρόπο σφαγή. Είναι απαράδεκτο οι καταναλωτέ να είναι υποχρεωμένοι να ε, αγοράζουν κρέα που έχουν, έχει, από ζώα που έχουν σφαγεί με τρόπο που δεν έχουν επιλέξει. Και πολλές φορές να βρίσκονται προϊόντα κατάλληλα στο κανονικό δίκτυο διανομής. Όπως οι καταναλωτές για προσωπικούς τους λόγους θέλουν να μπορούν να καταδικάσουν ή όχι την σφαγή για θρησκευτικούς λόγους που κάνει τα ζώα όχι μόνο να υποφέρουν αλλά με την... με τον αποκεφαλισμό ε, ενώ το ζώο ε, βρίσκεται σε ζωή προκειμένου να υπάρχει ανάλογη ροή αίματος ε, που δεν θα αλλάξει την ποιότητα του κρέατος, αυτά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά να φαίνονται στην επισήμανση, τη σωστή επισήμανση των προϊόντων κρέατος για την ε, σωστή ενημερώση των καταναλωτών. Ευχαριστούμε ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ενώ συζητούμε για ένα έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο νομίζω «Υλοποίηση του κανονισμού για τα σφαγεία», ε, πιστεύω ότι τελικά πέραν από το έγγραφο βλέπουμε μια δραματική εικόνα των δημοσίων σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι εδώ δεν βλέπουμε τι εικόνε των ζώων ε, που περιμένει κανεί να, να συναντήσει σε ένα σφαγείο. Βλέπουμε ένα σκύλο, ένα γατί, ένα άλογο και μια γελάδα. Σε κάποιε χώρε τη Ευρώπη όντω μπορεί να υπάρχουν γατιά και σκύλοι σε σφαγεία, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση θα το βρει κανεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν λοιπόν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την παίρνουμε σοβαρά, θα έλεγα τουλάχιστον να αλλάξουν την εικόνα στο εξώφυλλο αυτού του εγγράφου διότι η παρουσίαση ανέφερε επιπλέον και επιθεωρητές στα σφαγεία. Ε, έχω κάθε κατανόηση για όσους είναι υπεύθυνοι για τα βρετανικά σφαγεία που μπορεί να προέρχονται από χώρα όπου η θανάτωση αλόγων και τάβρων γίνεται για σκοπούς ε, θεάματος. Όμως αυτό παρόλο που με λυπεί ε, δεν πάβει να σημαίνει ότι ο Βρετανός φορολογούμενος ε, χρηματοδοτεί αυτές τις δραστηριότητες των ελεγκτών με τις χώρες που έρχονται από εκεί που οργανώνονται τα προμαχίες, οι υποδρομίες. Πάντως βλέπω ότι ως προς τη σφαγή των ζώων αυτό που θυμώνει τους Βρετανούς καταναλωτές είναι ότι δεν υπάρχει σαφής ετικετοθεσία, σαφής επισήμανση. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα μπορούσε να στιγματιστούν τα προϊόντα έτσι. Δεν με νοιάζει καθόλου προσωπικά. Ο καταναλωτή έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει όχι μόνο πώ έχει παραχθεί το προϊόν, αλλά και πώ θανατώθηκε το ζώο. Και όσο πιο ε, γρήγορα τα κράτη-μέλη αναλάβουν την αρμοδιότητα να βάζουν τι σωστέ ετικέτε, τόσο καλύτερα θα είναι, καλύτερα θα είναι οι πληροφορίε που έχουμε για τα προϊόντα μα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μίλναρ. Μάλιστα, Πρόεδρε. Έχουμε διαφορετικά προβλήματα εδώ ενώπιον μας. Αφενός έχουμε δυστυχώς μία επικέντρωση ότι τα σφαγεία έχουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις καλύπτουν μεταφερόμενα τα ζώα αυτά και είναι πολύ προβληματική η κατάσταση πόσο μεγάλες είναι οι αποστάσεις που καλύπτονται και υπό ποια πίεση βρίσκονται οι εργαζόμενοι στα σφαγεία στη συνέχεια. Αν αυτό τον κανονισμό τον κρίνουμε μετά από δύο χρόνια τον αποτιμήσουμε θα πρέπει να δούμε με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια αν αυτός ο κανονισμός είναι αποτελεσματικός ή όχι ή αν πρέπει να συμπληρωθεί και να βελτιωθεί. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια βελτίωση και ενδεχόμενα να υπάρξει ένα παράθυρο χρονικό για τη σφαγή των ζώων, είτε πρόκειται για βόηο κρέας, είτε χείριο, είτε πρόκειται για πουλερικά, είτε... Και ένα άλλο θέμα είναι το ότι αυτό το οποίο μας ε, με απασχολεί είναι, είμαι νέα σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και στην, βρίσκομαι στην διακομματική ομάδα Welfare Intergroup για την ευζοία των ζώων. Αν βλέπουμε τι γίνεται σε αυτά τα σφαγεία, ότι για παράδειγμα ένας τάβρος ε, προκειμένου να σκοτωθεί παλεύει, χαροπαλεύει 20 λεπτά μετά το χτύπημα που δέχεται, είναι απαράδεκτο αυτό. Πρέπει να ζητήσουμε στην Ευρώπη η ε, σφαγή χωρίς αναισθησία να μην επιτρέπεται πλέον. Πρέπει να τα ζώα και μετά να σφάζονται. Κατά πόσον λοιπόν μπορεί να βελτιωθεί αυτός ο κανονισμός ή βλέπει η Επιτροπή να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα γίνουν για την ε, ιχνηλάτευση, για την ανείχνευση του κρέατος ε, και την πιστοποίησή τους. Πρέπει το κρέας με αυτόν τον τρόπο να πιστοποιείται και να ε, διαφοροποιείται από τα άλλα ώστε να μπορεί το κρέας, το ζώο αυτό να έχει υποστεί την κανονική σφαγή με αναισθησία. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν τέτοιες βελτιώσεις. Η προστασία και η ευζοία των ζώων πρέπει να είναι ανώτατη προτεραιότητα και πρέπει με θάρρος να κινηθούμε ώστε να δράσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Κάπως ε, με εκπλήσει και ε, εξοργίζομαι στο ότι η συζήτηση περιορίζεται μόνο στις θρησκευτικέ εξαιρέσεις και το ότι ε, γίνονται παράπονα για την μη αναισθησία των ζών σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν δει κανεί τι γίνεται πραγματικά πρέπει να δούμε τι γίνεται στα σφαγεία και τότε πραγματικά δεν αληθεύουν όλα αυτά. Δεν είναι τόσο δεδομένα για την αναισθησία. Αν δει κανεί και εξετάσει τους χείρους για παράδειγμα όπου ήθιστε να αισθητοποιούνται με διοξίδιο του άνθρακα, βλέπει κανείς ε, πόσο απελπιστική είναι η κατάσταση αυτών των ζώων. Συνεχίζουν να ζουν μετά την ε, σφαγή τους αυτά τα ζώα. Είναι απίστευτο. Και προσπαθούν να ξεφύγουν, το ένα ζώο ανεβαίνει πάνω στο άλλο, είναι μέθοδος λοιπόν σφαγής που δεν είναι αποτελεσματική. Θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλουμε να αποστείλουμε ένα μήνυμα, να δώσουμε κάποιο μήνυμα, πρέπει να πάψει αυτή η μέθοδος σφαγής. Η ΕΦΣΑ έχει δώσει εδώ και πολύ καιρό αυτά τα μηνύματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Η εισήγηση, η έκθεση, ε, καλά ακούστηκε το 2013 ή τουλάχιστον τέσσερα κράτη βρισκόντουσαν σε θέση να εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό. Δανία, Γερμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα γίνεται λόγος ότι 70% των σφαγών καλύπτονται με τον σωστό τρόπο, γίνονται με τον σωστό τρόπο. Αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο ακούσαμε. Απουσιάζει όμως το 30% ακόμα από αυτό το 70% για να είμαστε πλήρεις και να καλύψουμε το 100%. Έχουμε το πρόβλημα του διοξιδίου του άνθρακα με τους χείρους. Έχουμε το πρόβλημα με, την, το ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τα πουλερικά. Μετά από το χτύπημα που υφίστανται στους, ε, ε κυλιόμενους ε, ε, στις κυλιόμενες ζώνες, στα σφαγεία βρίσκονται ακόμα ζωντανά πουλερικά, ζωντανά ζώα. Κάτι πρέπει να γίνει να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Συνολικά έχουμε πολλά να κάνουμε με τα προβλήματα σε σχέση με αυτό το σύστημα. Έχουμε λοιπόν ζητήματα τα οποία τίθενται σε σχέση με τα σφαγεία είναι λοιπόν ε, μαζικής εφαρμογής σφαγή και πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτό βρίσκεται υπό έλεγχο όταν βρίσκεται σε μαζική κλίμακα αυτού του είδους η σφαγή και υπάρχει τέτοια πίεση όπως προαναφέρθηκε από συνάδελφο μετά από μεγάλες διαδρομές που καλύπτονται πρέπει νομοθετικά να καλύψουμε τα κενά. Εδώ έχουμε αξίες ευρωπαϊκές όπως την ευζοία των ζώων που πρέπει να διαφυλάξουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε με ένα τέτοιο σύστημα όταν πιέζει το σύστημα και η σφαγή δημιουργεί τεράστια ένταση, τεράστια πίεση και χωρίς επαρκή αναισθησία σφάζονται τα ζώα. Πρέπει σε βάθος να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με ένα τέτοιο κανονισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε τον λόγο κύριε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω προς τους κυρίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφενός είπατε ότι έχουμε ήδη καλή εφαρμογή σε σχέση με τη σφαγή όσον αφορά το ε, ερυθρό κρέας. Έμεσα είπατε ότι στο λευκό κρέας, στα πουλερικά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Θα ήθελα να επισέλθετε με περισσότερα στοιχεία και να αποσαφηνίσετε αυτόν τον τομέα που μεγεθύνεται και δεύτερον είπατε ότι η βιομηχανία, ένα συμβιβασμό μεταξύ ποιότητας λέει κρέατος και προστασίας των ζώων πρέπει να επιτύχει. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας. Διότι το υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων οδηγεί στην υψηλή ποιότητα του κρέατος. Και ζώα τα οποία σφάζονται χωρίς πίεση και χωρίς άγχος και με τις σωστές διαδικασίες οδηγούν σε αναβαθμισμένη ποιότητα κρέατος μετά τη σφαγή. Αυτά όλα να τα λάβετε υπόψη σε σχέση με τις τοποθετήσεις σας. Δηλαδή για τον συμβιβασμό αυτό μεταξύ ποιότητας κρέατος και τρόπου σφαγής. Και με εκπλήσει πρέπει να πω επιπλέον αυτά τα οποία είπατε, αυτό που είπατε. Κάτι άλλο ανέμενα. Ίσως οι προσδοκίες μου δεν ήταν οι σωστές. Ίσως οι δικές σας τοποθετήσεις δεν ήταν σωστές. Θα ήθελα να δούμε σήμερα σε ποιους τομείς δεν ευθυγραμμίζονται οι μέθοδοι που ακολουθούμε με τη σωστή σφαγή. Και συγκεκριμένα δεν θέλαμε σε σχέση με το τι γίνεται με τις διάφορες θρησκείες προσκαλέσαμε εσάς και όχι θρησκευτικούς εκπροσώπους εσάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας πείτε με ποιο τρόπο σφάζονται τα ζώα ώστε να δούμε σε σχέση με τις ε, διαφορετικές ε, σφαγές ε, ή μεθόδους σφαγής τι γίνεται ώστε οι μικρές εξαιρέσεις που μπορεί να υπάρξουν ώστε να δώσουμε κάποια περιθώρια να επανεξεταστούν και να υπάρξουν νέοι, νέοι περιορισμοί και νέα, ε, νέοι, ε, νέοι προσδιορισμοί για την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις ε, στον κανόνα και αυτό θέλουμε να εξετάσουμε. Υποστηρίζω τους προλαλήσαντες. Πουθενά δεν καθίσταται τόσο εξόφθαλμο ότι η βιομηχανία πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες διαδικασίες από ό,τι στη σφαγή. Πρέπει να αλλάξει η νοτροπία τους. Πρέπει να προσαρμοστεί η νοτροπία των βιομηχανικών αυτών τρόπων σφαγής. Δεν είναι καθόλου αδιάφορο αυτό. Είναι θέμα αξιοπρέπειας και ένα θέμα του ότι κατά τη σφαγή πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε ατομικά να σφάζονται τα ζώα και να μην είναι απλά και μόνο αντικείμενα τα οποία θεωρούμε ότι οδηγούνται προς σφαγή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Εκ παρακαλώ και πάλι. Έχετε τον λόγο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είναι σχεδόν φάρσα όταν οικονομικές πτυχές του θέματος τις εξισώνουμε με πτυχές ευζοίας των ζώων. Εδώ συσχετίζονται αυτά σε σχέση με την ηθική, η ηθική και την, ένα ηθικό πλαίσιο και να μην συγχαίουμε τα βιομηχανικά με την ηθική. Ερώτηση, τι σχεδιάζει να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα στη σφαγή, στην αναισθησία και μετέπειτα σφαγή των χείρων. Είναι χωρίς αμφιβολία το ότι η αναισθησία με διοξίδιο του άνθρακα οδηγεί σε περί σε υπερβολικό άγχος ε, ε, τα ζώα αυτά, πράγμα που είναι και περιττό κιόλα και περιτεύει. Έγινε λόγος για χείρους, έγινε λόγος, λόγος για αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται με τις εκατοντάδες χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια κουνέλια που σφάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αυτό ένα είδος ζώο, το κουνέλι, που είναι εξίσου ευαίσθητο όπως και άλλα ζώα. Ακούσαμε για πουλερικά. Έχουμε κάποιες προόδους που έχουν σημειωθεί σε σχέση με κάποιους τομείς. Ακόμα και για την κτηνοτροφία, αλλά για κουνέλια δεν έγινε λόγος. Και ίσως και μια τρίτη ερώτηση εδώ, την οποία τώρα ε, μόλις σκέφτηκα να διατυπώσω. Έχουμε σχετικά υψηλές προδιαγραφές για την προστασία των ζώων στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε όλοι ότι ένας μεγάλος αριθμός ζώων ζωντανά εκτός των συνόρων της Ευρώπης μεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο. Και ακριβώς στα όρια της Ευρώπης προς μια τρίτη χώρα τι γίνεται, δεν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και ο κύριος Βοτσεχόφσκι το ανέφερε. Μεγάλοι όγκοι, μεγάλη αριθμοί ζώων μεταφέρονται στην Εγγύς Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, ζωντανά, μεταφορές ζώντων ζώων. Φρικτή κατάσταση η κατάσταση των ζώων και οδηγούνται εκεί σε μετά την άφηξή τους σε σφαγή. Δεν πρέπει εδώ πάλι κάτι να γίνει από πλευράς μας. Δεν είναι λογικό και να λέμε ότι μόνο στην Ευρώπη μπορούν να προστατεύονται τα ζώα αυτά όταν είναι ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκής προέλευσης ζώα τα οποία οδηγούνται και εξάγονται σε άλλες χώρες και αυτά πρέπει να προστατεύονται κατά τη μεταφορά και άφηξή τους εκεί. <clears throat> Σας ευχαριστώ και εγώ Πρόεδρε. Αυτή την εισαγωγή σε σχέση με τον προλαλήσαντα πρέπει να τονίσω ότι είναι σημαντική υπόθεση για την ηθική και την ηθική διάσταση του θέματος. Πρέπει να επιβάλλουμε στην οικονομία και στη βιομηχανία αυτές τις αρχές. Δεν είναι δυνατόν να είναι προαιρετικής εφαρμογής όταν βλέπουμε ότι ε, δεν επιτρέπεται λέει να αναισθητοποιούνται τα ζώα και σφάζονται χωρίς αναισθησία και υπάρχουν μόνο πολύ λίγες εξαιρέσεις και η προλαλήσαντα ανέφερε κάτι το σημαντικό. Είπε ότι και όταν υπάρχουν θρησκευτικές αρχές ή θέματα θρησκευτικού τρόπου σφαγής πρέπει να μετεξελίξουμε κάποια πράγματα και στην, ε, στην ίδια την Ομοσπονδιακή Βουλή στη της Γερμανίας συζητήθηκαν τα θέματα αυτά και προτρέψαμε τους ε, θρησκευτικά υπεύθυνου να τοποθετηθούν και είδαμε ότι είχαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους σε σχέση με την αναισθησία των ζώων. Αν δηλαδή μπορούσαν να ανασφάζονται με ή χωρίς αναισθησία. Ενδιαφέρον αυτό και πρέπει να υπάρξει μια μετεξέλιξη των πραγμάτων και αναπροσαρμογή τους. Ερώτησή μου υπάρχει είναι δυνατόν και προσθέτω τη φωνή μου σε εκείνους που είπαν ότι η σφαγή χωρίς αναισθησία δεν πρέπει να επιτρέπεται. Είναι αδιάφορο υπό ποια ιδιότητα γίνεται το ένα ή το άλλο. Τι πιστεύει ο υπεύθυνο, ε, ποιο ποσοστό είναι εκείνο το οποίο ε, εφαρμόζεται σήμερα σε σχέση με, αυτή, με αυτόν τον τρόπο σφαγής. Και όταν έχουμε σφαγή με ιεροτελεστικό τρόπο ως ιεροτελεστία θρησκευτική και σε σχέση με τις εξαγωγές που αναφέρθηκε αλλά και άλλο ερώτημα εξάγουμε πολλές φορές ε, κρέας σφαγίων από την Ευρώπη προς τρίτα κράτη ε, ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι ή εξάγουμε ζωντανά ζώα τα οποία σφάζονται στην άφηξή τους και μάλιστα χωρίς αναισθησία και σε αγορές τρίτων χωρών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών τρίτων χωρών. Τι ακριβώς γίνεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσείς τώρα έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και εγώ μένω κάπως έκπληκτη πρέπει να πω με αυτή τη συζήτηση σήμερα και θα ήθελα να εκφράσω από πλευράς μου την άποψή μου, δεν είχα υπόψη να παρέμβω, όμως δεδομένων των παρεμβάσεων που έγιναν πρέπει και εγώ να πω την δική μου άποψη σε σχέση με τον κανονισμό που βρίσκεται εν ισχύ, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ε, εδώ και δύο χρόνια περίπου που ισχύει, συμφωνώ, υπάρχει υλοποίηση και ευθυγράμμιση κατά 70% αν κατάλαβα καλά από τις παρεμβάσεις που έγινε, ε, από την παρέμβαση που έγινε από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και γι' αυτό πιστεύω είναι λογικό. Είναι λογικό αυτό το οποίο γίνεται και βρίσκεται υπό εξέλιξη. Άλλο πράγμα τώρα είναι ότι σε κάποια μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι αρεστός αυτός ο κανονισμός. Όμως έχει εγκριθεί αυτός ο κανονισμός και είναι ένας καλός κανονισμός και παράγει μια, προκαλεί μια αλλαγή στην Ευρώπη. Αλλαγή στην Ευρώπη συνολικά όσον αφορά το σεβασμό της ευζοίας των ζώων. Και αυτό είναι κάτι θετικό, είναι κάτι καλό. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τι γινόταν πριν, τις αλλαγές δηλαδή που έγιναν σήμερα και είναι καλές και θετικές και επιπλέον πιστεύω και κάτι άλλο, ότι ο σεβασμός ε, που εγκρίθηκε σε σχέση με κάποιες ε, μορφές ιεροτελεστικής σφαγής ε, λόγω, λόγω θρησκευτικών λόγων είναι κάτι που στην Ευρώπη διατηρείται και θα θέλα εγώ να πω με κάθε σαφήνεια ότι δεν θεωρώ ότι αυτό σημαίνει να ξανανοίξουμε νέα συζήτηση επί του θέματος και να αμφισβητήσουμε τα πάντα. Ο κανονισμός είναι σωστός και λογικός. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα από την οποία ξεκινήσαμε οι διάφορες χώρες. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, την Ισπανία, όπου η κτηνοτροφική παραγωγή είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει μια μετατροπή, αλλαγή όσον αφορά τις σφαγές στα σφαγεία. Ο ρυθμός και οι αλλαγές είναι θετικές. Κατανοώ τις ευαισθησίες που λένε ότι πρέπει να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο. Το κατανοώ αυτό, αλλά τα πράγματα πρέπει να έχουν την τάξη τους. Και η τάξη τους είναι η ανησυχία, το μέλημα που πρέπει να έχουμε στην Ευρώπη πρώτα και κύρια για τους πρόσφυγες και τους ε, ε, μετανάστες και πρέπει να προσπαθήσουμε το 100% να πετύχουμε το στόχο για την ευζοία των ζώων. <clears throat> Όμως ο κύριος λόγος ε, είναι, πρέπει να είναι στην Επιτροπή μας ε, για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τις εργασίες μας ε. και ο στόχος μας είναι κυρίως η ευζοία των ζώων αλλά όχι πάνω από την ευημερία των ανθρώπων, των ατόμων. Να μην λοιπόν δημιουργήσουμε προτεραιότητες που θα αντιστρέφουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Έχουμε φτάσει λοιπόν στην... στο τέλος του καταλόγου των ομιλητών. Ξαντλήσαμε τον κατάλογο. Λοιπόν, για να ζητήσουμε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γκαβινέλη, να σχολιάσει όσα ελέγχθησαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για, την, ε, για το ενδιαφέρον τους και τις ερωτήσεις που έθεσαν. Άνοιξε όμως μια ευρύτατη συζήτηση έτσι που αγγίζει και θέματα που έχουν να κάνουν με τη Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων, τη συνθήκη, την ε, Άνεξη θρησκεία, δεν μπορώ εδώ να πάρω θέση σε τέτοια θέματα. Ε, ξεπερνούν το πεδίο των αρμοδιοτήτων μου. Οπότε, για τις τεχνικές άμεσες ερωτήσεις θα κοιτάξω να απαντήσω. Να πω ευθύ αμέσω για τον αριθμό των ζώων που σφαγιαζόνται χωρίς ανιστοποίηση στην Ευρώπη. Προς στιγμή δεν έχουμε νομική διάταξη που να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες. Δεν συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό. Τα δεδομένα που διαθέτουμε προκύπτουν από μελέτες, μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέσω τρίτων. Για να δώσω ένα είδο απάντηση για τα βοηθή με μια μελέτη του 2012 γίνεται λόγος για έναν αριθμό περίπου 8,5% του συνόλου των σφαγισμένων ζώων σε ένα χρόνο. 2 εκατομμύρια ε, βόδια και μοσχάρια που σφαγίζονται θυσίως δηλαδή. Για τα υπόλοιπα είδη δεν έχουμε ακριβή δεδομένα και για αυτόν τον λόγο ακριβώς αυτές τις μέρες όλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να υπάρξει συνεργασία για τη συγκέντρωση πληροφοριών από τα 28 κρατη ώστε να υπάρξει μια εκτίμηση τουλάχιστον των αριθμητικών δεδομένων και περιμένουμε τα πρώτα στοιχεία για τις αρχές του 2016. Σε ό,τι αφορά τη διάσταση των εξαγωγών των ζώων προς τρίτες χώρες, Η παρουσίαση αφορούσε τις σφαγές σε τρίτες χώρες που εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις σφαγές σε τρίτες χώρες και την κατανάλωση εκεί, προφανώς αυτά διέπονται από τον κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και δεν μπορεί καθόλου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει σε διμερείς επαφές για τα θέματα αυτά, για την προστασία των ζώων, την υγεία τους και με τον υπεύθυνο οργανισμό ΤΑΓΕΚΣ για την ενημέρωση των Ευρωπαίων Καταναλωτών οργανώθηκε ένα πειραματικό σεμινάριο για τους φαγείς χωρών προορισμού των κράτων αυτών για να βελτιωθούν οι επιστημονικές τους γνώσεις. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα αυτό και θα δούμε αν μπορούμε να επενδύσουμε περαιτέρω στο μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση για να βελτιώσουμε τα πράγματα. ως προς τις εξαγωγές και ερχόμαστε σε μια από τις ερωτήσει κλειδιά ως προς την ε, νομιμότητα του να σφαγιάζει κανείς ζώα χωρίς αναισθητοποίηση και για την εξαγωγή κρέατος από ζώα που δεν έχουν αναισθητοποιηθεί ο κανονισμός και είχε και έχει ως βασικό στόχο να συνδυάσει τις ε, απαιτήσει, του κανόνε προστασία των ζώων με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η εξαίρεση πρέπει να ε, ερμηνευθεί κατά τρόπο περιοριστικό. Είναι λοιπόν σαφέ, το είπε και ο νομοθέτη, δεν είναι δυνατό η εξαίρεση απλώς να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τον κανονισμό, οπότε κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμόζουν αναπερίπτωση την εξαίρεση βάσει μιας έκθεσης που λαμβάνει υπόψη αυτές τις παραμέτρους. Γι' αυτό εδώ μιλάμε και για τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων εν παραλίλω. Δεν έχουμε μια γενική απάντηση για το αν το να σφαγιάζει κανείς χωρίς αναισθητοποίηση για σκοπούς εξαγωγών είναι νόμιμο ή όχι, για τον εξή απλό λόγο. Αναπερίπτωση, κράτο μέλος προ κράτο μέλο πρέπει να αξιολογείται διαφορετικά η κατάσταση. Αυτό έχουν απαντήσει οι αρμόδιοι μας. Ως προς την επισήμανση της ετικέτας και μια ερώτηση που εν μέρη απαντά η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ για τη μελέτη που ζητήθηκε και από το Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε ένα δείγμα πολιτών και τεχνικών φορέων που καλύπτουν το 80% της ευρωπαϊκής παραγωγής ως προς τις σφαγές. Υπάρχει και μια σχετική δημοσκόπηση με τη συμμετοχή Ευρωπαίων καταναλωτών και πολιτών από 28 ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε και είναι η πρώτη δεν δείχνει να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ να έχουν αυτέ τι πληροφορίε στην ετικέτα. Αυτό προκύπτει τη συγκεκριμένη μελέτη. Στι περισσότερε περιπτώσει υπάρχουν μάλιστα σαφεί απαντήσει από τη δημοσκόπηση που έγινε και όπω είπα αυτά διατίθενται και στο διαδίκτυο φαίνεται να μην μπορεί ο μέσος καταναλωτής να αξιοποιήσει την πληροφορία αυτή, διότι δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες με την ε, διαδικασία σφαγής. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή, ο καταναλωτής απαραίτητος τι θα πει αναισθητοποίηση. Στη μελέτη λοιπόν αυτή σίγουρα υπάρχουν ε, μέρημνες από πλευρές καταναλωτών για την προστασία των ζώων, αλλά δεν είναι σαφές ότι η επισήμανση είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχουν τις πληροφορίες αυτές στα χέρια τους. Το θέμα αυτό πρέπει να το μελετήσουμε, σαφώς το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για αυτό το σκοπό ε, μια μελέτη για τις γενικές πληροφορίες που προσφέρονται στους Ευρωπαίους καταναλωτές για την προστασία των ζώων θα δημοσιευτεί και κατά πάσα πιθανότητα το σύνολο των στοιχείων θα ε, αξιοποιηθεί για να εκπονηθεί, να σχεδιαστεί μια σχετική στρατηγική. Σε ό,τι αφορά τον τεχνικότερο, το τεχνικότερο θέμα για τους πειραματισμούς και τη χρήση διοξιδίου του άνθρακα στο, στην αισθητοποίηση. Να το πω ευθύ αμέσως. Όταν είπα συμβασμό εξισορρόπηση μεταξύ ποιότητα και προστασία των ζώων, δεν εννοώ ότι η υγεία των ζώων βλάπτει την ποιότητα του κρέατο, ε, του αντίον. Τον προστατεύει κανεί επαρκώ τα ζώα από την πρώτη μέρα ζωή του είναι ένα καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα του τελικού προϊόντο και εκτιμάται δεόντω. Σε ό,τι αφορά όμω την ανεξιτοποίηση των ζώων, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη τεχνολογική ε, φάση εδώ. Η αρχή για την επιστημιστική ασφάλεια και για του χείρου και για τα πολιτικά έχει επισημάνει ότι το σύστημα του διοξιδίου του άνθρακα δεν είναι μεν τέλειο, αλλά είναι αποτελεσματικό για να μπορέσει να υπάρξει απαραίτητη ποιότητα για την ε, υγεία των ζώων. Ταυτόχρονα όμως η ανάλυση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό ε, Εμπορικό Σύστημα δεν επέτρεψε να διαφανούν βιώσιμες εναλλακτικέ για τον ευρωπαϊκό κλάδο σε αυτή τη φάση. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή δεν ε, επέβαλε την ε, μετατόπιση από το, σύστη, το ηλεκτρικό σύστημα στο σύστημα διοξιδίου του άνθρακα για τα πουλαρικά, γιατί δεν υπήρχαν και ε, ε, δεν υπήρχε απαραίτητη προετοιμασία βραχυπρόθεσμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσει ανάλογε επενδύσει καινοτόμε και στην τεχνολογία για το θέμα αυτό, θα πρέπει να έχει τι ανάλογε αποδείξει στα χέρια τη. Και του κύριο ισχύει κάτι παρόμοιο με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή για τους χείρους το διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και με άλλα αέρια. Η κατάσταση λοιπόν σε γενικές γραμμές είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη. Όπως υπόθηκε, ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περνάει σε μια φάση εκκίνησης νέων στρατηγικών, νέων πολιτικών για το μέλλον. Οπότε οι πληροφορίες αυτές σαφώς είναι σημαντικότατες για να σχεδιάσουμε σωστά την μελλοντική μας προσέγγιση για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Όταν ξεκινήσαμε να συζητούμε αυτό το θέμα, είπα ότι ε, τα περαιτέρω βήματα θα πρέπει να αποφασιστούν αφού ακούσουμε τα σχόλια σήμερα. Λοιπόν, τι προτείνω. Προτείνω να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα στις ε, συναντήσεις συγκεκριμένων πολιτικών ομάδων, στις ομάδες δηλαδή, και αφού συζητηθεί το θέμα οι συντονιστές μπορούν να επιστρέψουν με τις απόψεις από τις πολιτικές ομάδες να μας φέρουν τις απόψεις στην συνεδρίαση των συντονιστών και εκεί να εξετάσουμε ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα. Όπως είπα, είναι μια πρωτοβουλία του ECR. Ε, ένα συγκεκριμένο σχήμα προτάθηκε από τους συντονιστές. Νομίζω ότι είναι σωστό προς το παρόν. Ας μην επιταχύνουμε χωρίς λόγο για να μην οδηγηθούμε σε ανεφλόγου εντάσεις ή συζητήσεις. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Έχει να κάνει με την ηθική. Λοιπόν, αυτό σας προτείνω για τα μελλοντικά βήματα επί του θέματος. Τώρα, έληξε η συνεδρίαση για σήμερα. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο το πρωί ψηφίζουμε. Σας παρακαλώ μην ξεχάσετε τη σχετική ηλεκτρονική κάρτα σας. Ο κύριος Άντρου θα προεδρεύσει αύριο, διότι υπάρχει μία συνάντηση υπουργών του Συμβουλίου αύριο στο Λουξέμβουργο. Ο κύριος Άνιου έχει το λόγο. Μπορεί να υπάρξει κάποιο μπέρδεμα κύριε Πρόεδρε τουλάχιστον στα αγγλικά. Είπατε ότι ο κύριος Άγνιου θα προεδρεύσει τη συνεδρίαση αύριο. Σας διαβεβαιώ πως δεν θα προεδρεύσω. Λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι παρόν, πρέπει να πάω σε μια κηδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρος. Ε, λάθος δικό μου λέει ο πρόεδρος. Κοιτούσα εσάς και δεν έβλεπα τον κύριο Άντριου που είναι απόν σήμερα. Άντριου λοιπόν. Άντριο μάλλον, για να το προφέρουμε και σωστά. Οκ, λοιπόν, αυτό θα προεδρεύσει αύριο και σε πέντε λεπτά θα έχουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ.